πλέον η ώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πάρει τα ενία στα χέρια του και να ε, υπερασπιστεί μόνο του την κοινοτική μέθοδο. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Πολύ καλά. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση. Ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Σούλτ. Επόμενο θέμα. ψήφιση με την απλουστευμένη διαδικασία της έκθεσης κυρίας Ματέρα. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Τομείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Ψηφίζουμε. Ονομαστικά. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια κυρία Ματέρα. Επόμενη έκθεση. Προβέρα μεταναστευτικά ρεύματα που οφείλονται στην αστάθεια. Πεδίο εφαρμογή και ρόλο εξωτερική πολιτική ένωση. Ψηφίζουμε. Ψήφι υπέρ είναι ενιαία η ψηφοφόρη. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ κύριε Προβέρα. Ερχόμαστε τώρα στην έκθεση Γέγκλε. Ο ρόλο των γυναικών στον τομέα τη γεωργία και στι αγροτικέ περιοχέ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Γέγκλε. Και τώρα έκθεση Μαρινέσκου. Χρηματοδότηση ένωση στο τομέα του παροπλισμού πυρηνικό σταθμό στα νέα κράτη-μέλη. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Μαρινέσκου. Επανερχόμαστε στην κυρία Ματέρα. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Τσεχική Δημοκρατία. Μία τροπολογία έχουμε εδώ. Γιατί ψηφίζουμε. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Παρακαλώ ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία παριθμών 1. Πέρασε. Εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε το σχέδιο ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική κλίση. Αρχίζει τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Ματέρα. Ερχόμαστε στην έκθεση Λάχισπριτ. Εξαγωγές ειδών και τεχνολογίες διπλής χρήσης. Έχουμε πολλές τροπολογίες. Ψηφίζουμε την 36 ψήφι υπέρ είναι της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Κατά. Αποχές εγκρίνεται εγκρίνονται, συγγνώμη, και οι 36 τροπολογίες της Επιτροπής. Η τροπολογία 8. Τσίφι Π. Κατά. Αποχές. Έλεγχο παρακαλώ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 8. Πέρασε. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 12 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Παρακαλώ για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 12. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία παριθμό 13 σε τρία τμήματα. Τμήμα πρώτο ψήφι Π. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τμήμα δεύτερο ψήφι Π. Κατά. Αποχές έλεγχος παρακαλώ. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας υπαριθμών 13. Check is... Πέρασα. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Ψήφι Π. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21 ψηφίπε Κατά. Αποχές. Ε, ε, έλεγχος παρακαλώ ηλεκτρονικός για την 21. Άρχεται. Πέρας τώρα. Εγκρίνεται. Η τροπολογία παριθμό 38 ψήφι Κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχο θέλετε. Καλώς. Άρχεται. Ο έλεγχος για την 38. Πέρας. Απορρίπτεται. Όντως. Η 44 ψήφι πέρα. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί, αλλά στην ελέγξουμε καλύτερα. Την 44 παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε. 23 ψήφι Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ε, σας ζητώ συγγνώμη. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 23. Check is Πέρας. Ε, απορρίπτεται. 48 ψήφι πέρα κατά αποχές απορρίπτεται. Και εδώ έλεγχο θέλετε, γιατί 48 αρχίζει τώρα ο έλεγχος. Πέρας. Εγκρίθηκε. Ζητώ συγγνώμη. 33 ε, ψήφι πέρα. Κατά. Αποχές Ελέγχεται παρακαλώ 33 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Έχω αρχίσει να κλονίζομαι. Check is closed. Πέρασε. Α, απορρίφθηκε. Σαραντανέα. ψήφιπε Κατά. Αποχές. απορρίφθηκε Έλεγχο. Αρχίζει η ψηφοφορία για τις 49. Πέρας της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Ζητώ συγγνώμη και πάλι. Και ερχόμαστε στην τροπολογία 42 ψηφιπέ. Κατά. Αποχές. Ας το ελέγξουμε. Εγώ νομίζω ότι απορρίφθηκε, αλλά ας το ελέγξουμε. Αρχίζει τώρα για τη 42 ηλεκτρονική υπολήθευση. Πέρας. Απορρίφθηκε όντως. Και ερχόμαστε στην τροπολογία υπαριθμό 50 ψήφι πέρα Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχο. Έλεγχο. Γιατί 50 αρχίζει ηλεκτρονική παλήθευση. Πέρας. Adopted. Εγκρίθηκε. 46 ψήφι πέ. Κατά. Αποχές. Ας την ελέγξουμε και αυτή. 46. Αρχίζει η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Δεν ξέρει κανείς ποτέ. Απορρίφτεται. 51 ψήφι Κατά. Δεν είναι σαφές. Ζητώ συγγνώμη. Ε, ελέγχουμε και την 51. Αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική πολίθευση. Πέρας. Εγκρίνεται. 47 ψήφι Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Γιατί 47. Πέρας. Απορρίπτεται. Η πρόταση της Επιτροπής, όπως ε, τροποποιήθηκε, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή για ένα διαδικαστικό ζήτημα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας οδήγησε σε κάτι που μπορεί να είναι συζητήσιμο επί της ουσίας, αλλά είναι πολύ κοντά στη θέση του Συμβουλίου πλέον. Και θα ζητούσα με τους σκιώδεις συγητές να αναβληθεί η τελική ψηφοφορία. Γιατί είναι πολύ μεγάλη πιθανότητα τελικά να επιτύχουμε συμφωνία με το Συμβούλιο. Θέλει να πει τίποτε Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι, μιλάει στο τηλέφωνο, στο iPhone, λέει ο πρόεδρος. Right. Well, in the absence of a commission opinion... ε, απουσία της Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Ποιος είναι υπέρ τη αναβολή τη τελικής ψηφοφορία. Παρακαλώ. Κατά. Αποχέ. Ούτως και αναβάλλεται. Ευχαριστώ κύριε Λάιξφριτ. Πολύ καλή δουλειά. Έκθεση του κυρίου Ζαντό εξαγωγικές πιστώσεις που την χάνουν δημόσια στήριξη. 21 τροπολογίες μαζί όλες, ψήφι υπέρ της Επιτροπής Εξωτερικού Εμπορίου, κατά, αποχές εγκρίνονται. Ποιος θέλει το λόγο? Ο κύριος Σόλτς. Όχι ο κύριος Σούλτς, ο κύριος Σόλτς είπα. Μάλιστα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ανακοινώσω ότι θέλω να αποσύρω εξ ονόματο τη ομάδα μου της ενωτική Αριστεράς την ονομαστική ψηφοφορία που έχουμε ζητήσει στην τροπολογία 10 και στα δύο τμήματα αυτής. Καλώ. Ψηφίζουμε τη 10 λοιπόν σε δύο τμήματα. Ψήφι υπέρ του πρώτου. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα είπε κατά, αποχές, έλεγχος. Λυπάμαι, απέσυρε την ονομαστική ψηφοφορία, γι' αυτό τώρα το λέω. Το δεύτερο τμήμα. Πέρασε. Εγκρίνεται. 22 ψήφοι πέ, κατά αποχές Νομίζω ότι απερίφθη, αλλά στην ελέγξουμε καλύτερα. 22 ηλεκτρονικά. Αρχίζει η παλήθευση. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Η πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Κύριε Ζαντό, έχετε το λόγο. Monsieur le Président, euh, Ευχαριστώ πολύ. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, οι σκιώδεις και ο υποφαινόμενος ζητάμε να μην ψηφιστεί από την Ολομέλεια για να συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, ελπίζοντας πως θα λάβει υπόψη τα όσα ψηφίστηκαν σήμερα εδώ στο Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε το λόγο. Έχετε το λόγο. Δεν θέλει να μιλήσει ο Επίτροπος. We Ψηφίζουμε την αίτηση ε, αναβολής Είπε κατά αποχές. Αναβάλλεται λοιπόν η τελική ψηφοφορία. Επόμενο και τελευταίο θέμα για σήμερα το πρωί είναι η έκθεση κυρία Φένσον πλαίσιο πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Παράγραφος 2. Αιτιολογική αναφορά 1 με ονομαστική κλίση. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Παράγραφος 2. Αιτιολογική αναφορά 4 και πάλι ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται επίση. Παράγραφος 2, αιτιολογική αναφορά 10. Ψήφι Κατά. Εγκρίνεται. Παράγραφος 2, αιτιολογική αναφορά 11. Ψήφι Κατά. Αποχές έλεγχος. Παράγραφος 2, αιτιολογική αναφορά 11. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Παράγραφος 2, λογική αναφορά 12, ονομαστικά αρχίζει τώρα. Πέρασε. Εγκρίνεται. Παράγραφος 2, αιτιολογική αναφορά 14 σε δύο τμήματα και ονομαστική κλίση. Πρώτο τμήμα τώρα. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα, ονομαστικά, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρασε. Απερίφθη. Παράγραφος 2, τεολογική φορά 19. Με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Παράγραφος 7. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία ονομαστικά. The vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19 τμήματικά. Το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα της 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 ονομαστικά ξεκινάει η Λίγη. Εγκρίνεται. 28 ονομαστικά και πάλι ξεκινάει. Λίγη. Εγκρίνεται. 29 ονομαστικά ξεκινάει. Λίγη. Εγκρίνεται. Εκτιμώντας J σε τέσσερα τμήματα. Το πρώτο τμήμα από τα τέσσερα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Επαλήθευση για το τρίτο τμήμα του J, Ξεκινάει. Λίγη. Εγκρίνεται. Το τέταρτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ωραία. Ε, ας το υπεληθεύσουμε Για το τέταρτο τμήμα ξεκινάει η ηλεκτρονική επαλήθευση. Λίγη. Εγκρίνεται. Όμικρον, ονομαστικά, ξεκινάει. Λίγη. Ωραία. Όλο το ψήφισμα μαζί λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ωραία λοιπόν, τελείωσαν οι ψηφοφορίες. Ε, συγχαρητήρια στην κυρία Σβένσον και καλή όρεξη σε όλους τους υπολείπους.